Ξεκινάμε. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε, έχουμε πολλές ψηφοφορίες και ο κόσμος ταξιδεύει την Πέμπτη, οπότε καλό είναι να ξεκινάμε. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Για τα γλωσσικά σημειώστε δανέζικα, κροατικά και ελλανδικά δεν υπάρχουν σήμερα. Κάτι άλλο τεχνικό από τις τεχνικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμε αυτή τη μεγάλη αίθουσα συχνά και όταν μιλάτε επειδή είμαστε λίμπε και χρησιμοποιούμε αυτή την αίθουσα ε, πρέπει να έρχεστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί οι διερμηνείς ε, δεν μπορούν να σας ακούσουν αλλιώς απλά σας το διαβιβάζω γιατί κάποιοι συνάδελφοι μιλάνε μακριά από το μικρόφωνο Οπότε, η ψηφορία του κυρίου Νάγκη θα είναι 40 λεπτά, οι άλλες θα είναι πιο σύντομες, έτσι για να έχετε μία ιδέα. Πριν πάμε στις ε, ψηφοφορίες, έχουμε το σημείο 3 των πρακτικών της συνεδρίασης ε, της 3 Οκτωβρίου 31 Αυγούστου και 30 ε, Μαΐου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Περνάμε λοιπόν τώρα στην πρώτη ψηφοφορία που είναι αυτή εδώ σημείο 5 έχουν όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες ε, ψηφοφορίας αλλιώς να το πούν τώρα. Ωραία, έχουμε όλες τις κάρτες. Σημείο 5. Σημείο 4. Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γεωργίας και Ευρωπόλ. Ο εισηγητής είμαι εγώ. Πάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τραπολογία 3. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Και αυτή απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ναι, 31 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 6 εποχές. Σημείο 5 για την Συμφωνία για Επιχειρησιακή και Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Europol. Η κυρία Γκαμπριέλ είναι η συγγήτρια. Περνάμε στην ψηφοφορία. Και αν συμφωνείτε μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες μαζί, 1 έως 4, ναι. Δεν θέλετε. Καλώς. Τροπολογία 1 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Έχει τελειώσει η ψηφοφορία και απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται τροπολογία 4 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται και αυτή. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 34 υπέρ 3 κατά 6 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στο σημείο 6, το μέσο ευελιξίας για μέσα του προπολογισμού για την συνεχιζόμενη κρίση προσφύγων και μεταναστών. Η συγκεκριά κυρία Μακοβέη. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική τέσσερα άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δέκτη τελική ψηφοφορία στο κείμενο που τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 38 υπέρ 3 κατά 2 αποχές συγχαρητήρια και περνάμε στο σημείο 7 το κινητοποίηση του αποθεματικού ανάγκης. Πάλι κυρία Μακοβέη, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική 1, άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτέ. Συμβιβαστική 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 21 άρχεται. Πέρας. Τροπολογία 22 άρχεται η ψηφοφορία. Είχε απορριφθεί η προηγούμενη. 22 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας δεκτή συμβαστική 4 αρχιτή ψηφοφορία πέρας δεκτή και το κείμενο όπως τροποποιήθηκε αρχιτή ψηφοφορία πέρας δεκτή 38 υπέρ 3 κατά 3 αποχές συγχαρητήρια στην εισηγήτρια σημείο 7 8 ε, στο σημείο 8 η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015 συγχύσω ο κύριος Νάγκη να αναφέρω κάποιες διορθώσεις στον κατάλογο ψηφοφορίας μετά από τις τροπολογίες 587 και 610 θα ψηφιστούν χωριστά γιατί το κείμενο έχει επαναλήψει σε περίπτωση περάσει η 587 θα καταπέσει 610 το ίδιο και με τις 702 953 οπότε αν περάσει 702 η 953 καταπίπτει. Αν το καταλάβατε όλοι, προχωράμε. Και να πω σύντομα, ο εισηγητής θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες, όλους τους κοιόδης και όλους τους βουλευτές για την τεράστια δουλειά πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Χίλιες τροπολογίες σχεδόν είχαμε. Καλύπτονται ε, όλες, 45 συμβαστικές έχουμε και μόνο 42 χωριστές ε, ψηφοφορίες. Ε, πολύ καλή δουλειά. Νομίζω πως η έκθεση αυτή θα δείξει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συνεργαστεί και να βρει ε, λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νάγκη. Περνάμε στην ψηφοφορία συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, δεκτή συμβιβαστική 3. 3 μέρος πρώτο αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 2.92 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 309 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4, μέρος 1, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Μέρος 2, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 8, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβεστική 37 μέρος πρώτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας δεκτή συμβιβαστική 6 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή τροπολογία 372 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 31 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 7. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, θα... Ε, δεν ξέρω αν καθίστε κάπου αλλού. Δεκτή. Καταγράφεται η ψήφος κ. Μπέκερ. Τροπολογία 404. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 406. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 αρχιετη ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Τροπολογία 416 16. η ψηφοφορία. Πέρας. Συμβαστική 11 αρχιετή ψηφοφορία. πέρας δεκτή 441 άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Συμβιβαστική 12 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 40 Άρχιτη ψηφοφορία. πέρας αδεκτή συμβαστική 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή συμβαστική 14 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή συμβαστική 19 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Ε, τροπολογία 487 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 16. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 17. Άρχεται ψηφοφορία. Δεκτή. Ε, πέρας. Δεκτή. 5.05. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5, 7, 8 και 5, 7, 9. Πανομοιότυπες άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 23. Με συγχωρείτε συνάδελφοι, 580. Άρχεται η συγχωρία. Ναι, 580. 580. ξανά παντε Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, με συγχωρείτε. Πρώτο τμήμα. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 587. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. συμβεστική 21. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 610. Όχι, πάμε στην 613. Άρχεται η ψηφοφορία. 613. πέρας Απορρίπτεται. 614. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν Εγκρίνεται. 694. άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Δεν Εγκρίνεται. 702. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Άρχεται το ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται το ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται το ψηφορία. Πέρας. Συμβαστική 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμ... Τροπολογία 738. Ναι, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβαστική 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 757. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 758 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 771 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38. Άρχεται η Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβαστική 38. Άρχιτη ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, ναι, μόλις κάναμε τα διδόκτω. 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 931. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 945. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 951. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 952. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 956. Τροπολογία 956. 953 καταπίπτει. 956. 956 Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 959. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 973. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, θέλετε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. 973 έως 982. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. Συνάδελφοι, αιτιολογικές αναφορές. Έχουμε ψηφίσει 7. Θα είμαστε στη σελίδα 55. Τροπολογία 1. Συνάδελφοι, τώρα θα ψηφίσουμε τις συμβαστικές προτάσεις για τις ιδεολογικές αναφορές. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστικό κείμενο για τις ιδεολογικές αναφορές. Πέρας. Εγκρίνεται. Εφόσον εγκρίνεται λοιπόν, πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Έτοιμε για τις αιτιολογικές σκέψεις. Πάμε απευθεία στο 118. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 118. Στις αιτιολογικές σκέψεις το βρήκατε όλοι. Πάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τα έχετε βρει όλοι. Ωραία. Συμβαστική 10 από τις, συμβαστικές σκέψεις, από τις αιτιολογικές σκέψεις. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 165. Αιτιολογικές σκέψεις. Άρχιτε ψηφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Τροπολογία 184 αιτιολογικός καψιών. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 254, 254, η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 260. Άρχιτε, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 270. Άρχιτε, η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα Πάμε στι παραγράφου τη Επιτροπής ΦΑΜ 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Επιτροπή Γυναικών ΦΑΜ 6. Άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. ΦΑΜ 56 έρχεται η ψηφοφορία. ΦΑΜ 56 πέρας. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι, τελική ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν άπαντε στην τελική ψηφοφορία. Όλοι ψήφισαν. Πέρα. Εγκρίνεται. 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 4 αποχέ. Συγχαρητήρια στον κύριο Νάγκη. Μπράβο σα. Τώρα να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Έχουμε άλλε δύο. οι κανόνες αστικού δικαίου για τη ρομποτική συντάκτη νομοδότησης ε, Μιχάλ Μπόνι. Έγκριση του σχεδίου νομοδότησης. Κύριε Μπόνι, θέλετε να πείτε τίποτα. Αν όχι, μπορούμε να αρχίσουμε τη ψηφοφορία. Οπότε. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 άρχεται. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική 10 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Συμβαστική 14 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Τώρα περνάμε λοιπόν στις αιτιολογικές σκέψεις. Α, συγγνώμη, τροπολογία 79 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Α, να περάσουμε στο 87. 87. 87 παρακαλώ. 87 Σωστό έτσι. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα, αιτιολογικές αναφορές και σκέψεις. Συμβαστική 1 για τις αιτιολογικές σκέψεις άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Και η τελική ψηφοφορία επί του κειμένου άρχεται. Πέρας εγκρίνεται 4702 συγχαρητήρια στον κύριο Μπόνι ευχαριστώ Τόμας αυτό μας βοηθάει ιδιαίτερα συμφωνώ αλλά εν περιπτώσει δεν πειράζει και τώρα έχουμε και μια άλλη έκθεση Μπόνι 10 Ανταλλαγή προφοριών, σύστημα έγκυρες προειδοποίησης για διάφορες ψυχοενεργές ουσίες. Και πάλι εισηγητής ο κύριος Μπόνη. Ψηφίζουμε για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και για τη της, ε, την ε, σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Εάν ο εισηγητής δεν θέλει να πάρει το λόγο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία. Δεν θέλει να πάρει το λόγο. Ωραία. Ωραία. 10 άρχεται. Πέρας. Δίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενδυ 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Στροπολογία 27 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένβι 14 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. MV15 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. MV16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. NV17 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Είναι ταυτόσιμη με το 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένβη 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 34, τέσσερα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμβη 23 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμβη 24. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμβη 25. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμβη 26. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές ε, σκέψεις. NV1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, καλή προσπάθεια. NV2. NV2. NV2. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. NV3. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. NV4. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. MV5 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. NV6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμβι 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμβι 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε η τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, 3 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε την απόφαση για να δώσουμε εντολή και για τη σύνθεση της διαπραγματευτικής μας αντιπροσωπείας. Άρχεται. Εντολή για ένεξη διαπραγματεύσεων. Πέρας. 48 υπέρ, μία ψήφος κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπόνι. Λοιπόν, τώρα έχουμε το 11. Είναι η ερώτηση, η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τις υποχρεώσεις της στον τομέα της αμοιβαιότητας των προξενικών θεωρήσεων με βάση το άρθρο 1.4 του κανονισμού 539.01. Είναι μία ενιαία ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 45 υπέρ, 3 κατά, 4 εποχές. Οπότε έληξε ο χρόνος ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας και για την παρουσία σας. Λοιπόν, συνάδελφοι, ήταν πολύ ταχεία ψηφοφορία. Είμαστε λοιπόν μια ώρα. Έχουμε κερδίσει μια ώρα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε διακοπή για τη βοήθειά σας και θα διακόψουμε για μία ώρα.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 Thank Ευχαριστώ. Έλεγε το παιδί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

μια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

Uh, dear colleagues, if Συνάδελφοι, αν θέλετε να ξεκινήσουμε, να είστε εδώ, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πήγαμε στις προφορίες πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε και πάλι λοιπόν ευχαριστώ για τη συνεργασία και την υπομονή και ευχαριστώ που ήρθατε στην ώρα σας. Ξεκινάμε με το σημείο 12. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Νέφους έκθεση του κυρίου, ε, σχέδιο γνωμοδότηση με τον κύριο Μπόνη, ε, είναι αρμόδια η Επιτροπή Ήτρε. Η ΛΥΜΠΕ όμως θα γνωμοδοτήσει βάσει του άρθρου 53. Και μου θυμίζουν εδώ να εξηγήσω κάτι που δεν κάνω συνήθω, ότι έχουμε πολύ καλό ιστορικό στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Είχαμε την εξέταση για την μαζική παρακολούθηση που είχε σχέση με τα θέματα του νέφους και θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε τι αρμοδιότητε μα σε αυτόν τον τομέα. Ο κύριο Μπόνι είναι πραίων του χώρου και αυτό ακριβώ θα φανεί και με αυτή την έκθεση ξανά. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε το τι έχει να πει σχετικά και θα του ζητήσω να πάρει το λόγο για να μα παρουσιάσει την έκθεση του, την νομοδότησή του μάλλον. Έχετε το λόγο κύριε Μπόνι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, έχω ετοιμάσει ένα σχέδιο γνωμοδότηση όπου επικεντρώνομαι στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και στηρίζω την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ανοιχτού επιστημονικού νέφους που να συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και γι' αυτό επικεντρώνομαι στην προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Υπογραμμίζω πόσο σημαντικό είναι για τους επιστήμονες και τους ερευνητές να μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα διότι αυτό είναι θεμελιώδη καινοτομία. Οι νέε τεχνολογίε και οι λύσει που προσφέρουν, όπω ε, η υπολογιστική νεφου και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Ανοιχτού Νεφου, θα φέρουν θετικά αποτελέσματα για τι επιστημονικέ εξελίξει και την καλλιεργία τη καινοτομία. Η ανταλλαγή δεδομένων και η επεξεργασία του θα πρέπει να γίνεται σε συμμορφώση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ε, ιδιαίτερω με βάση τον κανονισμό, τον Γενικό Κανονισμό για τη Βασική Προστασία των Δεδομένων. Πρέπει να βεβαιωθούμε από τώρα ότι υπάρχει αναρμονισμένη προσέγγιση ω προ την υλοποίηση του GDPR, όπω λέγεται, και αυτό είναι ε, καθοριστική σημασία για την επιστημονική κοινότητα. Να υπάρχουν οι ίδιε υποχρεώσει και οι ίδιε αρχέ να διέπουν ε, όλο το σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, εφόσον στι χώρε μα ασχολούμαστε με το, θέμα, με το σκέλος της υλοποίηση. Έτσι, η εναρμόνιση θα πρέπει να παραμείνει βασικό στοιχείο του προτινόμενου κανονισμού. Επίσης, για τις ελεύθερες ροές δεδομένων, ε, και αυτό καλύπτεται στην έκθεση για την ανάπτυξη της έρευνας και της ε, επιστημονικής κυρίως έρευνας, και ελπίζουμε και αυτή η πτυχή να καλυφθεί από την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Νομίζω μάλιστα τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει κάτι σχετικό. Ε, και εν τέλει υπογραμμίζω την σημασία της κυβερνοασφάλειας για το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Ανικονέφος για να αποφύγουμε τις, ε, τα ρήγματα στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη επιστημονικών λύσεων που θα επιτρέψουν να ε, Παρέχεται ασφάλεια στην ανταλλαγή και την επεξεργασία δεδομένων. Συνάδελφοι, οι εισηγητέ αποφάσισαν να εργαστούμε μόνο στα αγγλικά για το θέμα αυτό, καθώ θα πρέπει να ψηφίσουμε ήδη το Δεκέμβριο και να ε, υιοθετήσουμε την γνωμοδότηση πριν την ψηφοφορία στην Ήτρε. Η προθεσμία την υποβολή τροπολογιών στα αγγλικά μόνο είναι Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στι 6 το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προβλέπεται τον Δεκέμβριο στις 8 του μήνα. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε το θέμα, να ανταλλάξουμε απόψεις και βεβαίως για να συνεργαστούμε στενά με όλους τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε κύριε Μπόνη. Να περάσουμε τώρα στους κοιόδης και στους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ε, για τη γνωμοδότηση αυτή, πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω το έργο του συναδέλφου, του κυρίου Μπόνη. Για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης. Να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τους στόχους του όλου τα τέσσερα σημεία δηλαδή, τα σημεία κλειδιά για το όλο ζήτημα. Είμαι ικανοποιημένη που μπορώ να ασχοληθώ με ένα τέτοιο είδους θέμα. Ένα θέμα πολλά υποσχόμενο, με ιδιαίτερη αξία ευρωπαϊκή και ε, γενετικό υλικό, θα έλεγα, ε, επιστημονικό, το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε δημιουργικοί και εφάνταστοι. Εδώ έχουμε να κάνουμε την ανταλλαγή γνώσεων, την πρόθεση της ανταγωνιστικότητας και την πρόοδο της ψηφιακής ε, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενότητα. Αυτό και το επόμενο σημείο, το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά, ευτυχώς δεν αφορά ένα τόσο τραγικό θέμα όπως ε, συχνά θέματα τέτοιου είδους απασχολούν την ε, Επιτροπή μας. Δεν είναι τραγικής διάστασης. Εδώ λοιπόν βρίσκονται υποσιακή την ποικιλομορφία των δεδομένων που διατίθεται προς ανταλλαγή και που συνυπάρχουν στον έφος, νέες ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων, για την έρευνα, και για την επεξεργασία και το σχεδιασμό των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών. Χαιρετίζω λοιπόν αυτήν την διάσταση ευθύ εξ αρχή. Είναι σημαντικό να μπορούμε όχι να βρεθούμε ούτε ουραγή, αλλά ούτε στο μέσο τη όλη προσπάθεια, αλλά ε, όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τις ΗΠΑ και την Ασία. Μέσα από την γνωμοδότηση αυτή μπορούμε να δείξουμε δρόμους για να αναπτυχθούν τα εργολεία μας, τα οποία θέλουμε να είναι ευρωπαϊκά. Πρόκειται για εξαιρετικό θέμα και σύνολο θεμάτων. Βεβαίως προκύπτουν κάποιες ε, προκλήσεις και δυσκολίες, οι οποίες σωστά έχουν εντοπιστεί ήδη στις συνεννοήσεις μας, όπως από τη μία η προστασία και από την άλλη η ασφάλεια, και σε ό,τι αφορά την πτυχή της ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτό συχνά και αναφέρεται στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από τους πολίτες ως ανησυχία τους. Ο συνάδελφός μας σωστά εμένει στο σημείο αυτό διότι το νέφος, άρα το μελλοντικό ευρωπαϊκό νέφος, θα πρέπει να λάβει υπόψη τους κανόνες της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπου μπορούν να προκύψουν ε, δυσκολίες. Το σύστημα Λίζα παλιότερα είχε εντοπίσει τουλάχιστον 30 κινδύνους που μπορεί να προκύψουν λόγω του νέφους. Θα πρέπει λοιπόν να, κάνουν, να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση ε, και την ανταλλαγή δεδομένων που ε, βρίσκονται σε αυτό το νέφος δεδομένα τα οποία θα πρέπει με το ορθό σύστημα να προστατεύονται και βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων προς την πρόσβαση, τη διάρκεια τήρησης, την συλλογή, δεν θα δείξω τώρα της της ε, επιμέρους πτυχές, θα πρέπει να διασφαλίζονται. Δεύτερο σημείο που εγώ το θεωρώ άκρο σημαντικό είναι ο κίνδυνος τα δεδομένα που βρίσκονται σε ένα σύστημα ψηφιακό να αλλοιώνονται, να τροποποιούνται. Δηλαδή, ε, εναγνία των πολιτών να μεταβάλλονται ή ακόμα χειρότερα να επιτρέπεται πρόσβαση σε τρίτους, τρίτους οι οποίοι δεν έχουν τέτοια έγκριση, τέτοια άδεια. Λόγου χάρη, λόγω κάποιας ανεπάρκειας του συστήματος του παρόχου, ε, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που είναι παροχός ή λόγω κακοχρησίας από αυτόν τον ε, πάροχο, πέρα των τεχνικών ελλείψεων μπορεί να προκύψει μια τέτοια αλλίωση. Είναι σημαντικό η πτυχή αυτή να έχει ληφθεί υπόψη εξ αρχή και εκεί να προσφέρουμε τι απαραίτητε νομικέ εγγυήσει. Τρίτη υποσημείωση, αλλά και αυτή πολύ σημαντική, αφορά τις νομικές απαιτήσει για τα δεδομένα και τις νομικές, τις δικαστικές μάλλον ε, έρευνες που μπορεί να ζητούνται από τρίτα κράτη, από κράτη έξω ευρωπαϊκά. Αυτό είναι το πρώτο σύνολο θεμάτων που αφορούν την προστασία των δεδομένων και ως κοιόδης εντοπίζω και μια δεύτερη πρόκληση, αυτήν της ασφάλειας. Όταν ε, μιλάμε για το νέφος και τις ελευθερίες του, προκύπτει ένα μείζον πρόβλημα προστασίας δεδομένων που υπάρχουν στο νέφος, όπως είπα, έναντι της ε, κυβερνοασφάλειας, και του εγκλήματος των κυβερνοχώρων επιθέσεων που καταγράφονται και δημιουργούν δυσκολίες. Θα πρέπει με το κείμενό μας λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μία ε, επαρκή προστασία των υποδομών του μελλοντικού ευρωπαϊκού νέφους. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το δούμε από την αρχή, αντί να επιστρέφουμε και να αναζητούμε λύσεις στο θέμα όταν θα προκύπτουν τα προβλήματα μελλοντικά. Ως προς την ασφάλεια, η συγκέντρωση των δεδομένων είναι ένα δίκοπο μαχαίρι ως όπλο. Εκεί λοιπόν πρέπει να επιστήσω την προσοχή όχι μόνο στον εισηγητή που το γνωρίζει πολύ καλά, αλλά σε όλη μας την Επιτροπή και σίγουρα μέσα σε λίγε ώρε, γιατί προθεσμία νομίζω για την υποβολή τροπολογιών λείπει τη Δευτέρα, εδώ μέσα σε λίγε ώρε θα φροντίσω να υποβάλω σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νατάλη. Ο κύριος Αλιχά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω την άποψη του, του σκιώδους μας κυρίου Ντάλτον που δεν μπορεί να παρευρεθεί. Η γνωμοδότηση ε, φαίνεται εντάξει. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες αλλά θεωρούμε με ευχαρίστηση ότι πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Ντόλτον τονίζει ότι τον χαροποιεί ιδιαίτερα, ότι η γνωμοδότηση αναγνωρίζει ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων ήδη θέτει ένα ρωμαλαίο πλαίσιο. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω νομοθεσία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζούλη Σαχεντίνη. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος, ιδιαίτερα για επιστημονικούς σκοπούς, είναι πολύ καλή ιδέα. Υπενθυμίζω μια προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για παρόμοια πρωτοβουλία το 2013. 14, την περίοδο 13-14. Η Επίτροπος τότε, η Νέιλι Κρούς, είχε αρχίσει να αναπτύσσει το νέφος, αλλά επέλεξε δυστυχώς την Hewlett Packard για να εξελίξει το ευρωπαϊκό νέφος ενώ ήμασταν ε, σε φάση εξέτασης των αποκαλύψεων Σνόντεν. Εσείς ε, κύριε Πρόεδρε προεδρεύατε αυτής της ειδική Επιτροπής. Άρα υπήρχε θέμα προστασίας δεδομένων. Και είχαμε και τη δυνατότητα ε, να ευνοήσουμε κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες για να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό νέφος για να αξιοποιήσουμε τη δική μας περιοχή για να αποκτήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Για να δώσουμε τη δυνατότητα και στους Ευρωπαίους αλλά και σε άλλους να αποθηκεύσουν τα στοιχεία μας, τα στοιχεία τους σε εμάς. Και τι έκανε η Κομισιόν, επέλεξε τη Hewlett Packard και δεν έχουμε ακούσει και πολλά περαιτέρω. Καλό είναι που το συζητάμε όμως αυτό. Για να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία για να προστατεύει τους ε, Ευρωπαίους επιστήμονες και την εργασία τους. Εξετάζοντας τώρα την πρωτοβουλία, τονίζω ότι πρέπει να ευνοήσουμε τη δική μας, ε, το δικό μας κλάδο πληροφορικής και πρέπει να υπάρχει μεγάλη σημασία για την προστασία των δεδομένων. Οποιοδήποτε νέφος αποθηκεύει τέτοια ευαίσθητα δεδομένα δημιουργεί, δημιουργεί κίνδυνο για την ε, ιδιωτική ζωή των πολιτών και η Επιτροπή στην ε, ανακοίνωσή της το θεωρεί δευτερεύον. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες όταν ε, στέλνουν τα στοιχεία τους σε ένα τέτοιο νέφος. Πρέπει να το τονίσουμε. Ο, υπό το φως αυτής της σκέψης δεν συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η ψεύδο ανωνυμοποίηση και η ανωνυμοποίηση είναι ο σωστός τρόπος για να καλύψουμε το θέμα αυτό. Γιατί διαπιστώσαμε ότι μπορούν να αποκαλυφθούν εκ νέου τα πραγματικά στοιχεία. Δεν ε, καλύπτονται πραγματικά από την ψεύδο ανωνυμοποίηση. Δεν ξέρω αν είδατε την τελευταία εκπομπή Πανοράμα στη γερμανική τηλεόραση που έδειχνε τι μπορεί κανείς να μάθει για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι λοιπόν σωστός τρόπος η ανημοποίηση γιατί μπορούν να επανέλθουν εκ νέου στα αρχικά στοιχεία ορισμένοι. Επίσης θέλουμε να υπάρξουν προτάσεις και για υψηλού επίπεδου κρυπτογράφηση των στοιχείων. Ελπίζουμε λοιπόν η Επιτροπή μας να δώσει μια σωστή γνωμοδότηση και χαιρόμαστε για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τον κύριο Φως, αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Άξερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Εδώ η Επιτροπή μας εξετάζει το θέμα αυτό μόνο από πλευράς δικών μας αρμοδιοτήτων. Και πρέπει να τονίσω ότι στον ψηφιακό κόσμο ένα νέφος έχει διάφορες ε, πτυχές. Φυσικά τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να προστατεύονται τα δεδομένα. Αλλά αυτό σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει να προστατεύσουμε και την οικονομία μας, την ανταγωνιστικότητά μας υπάρχουν νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, μη επανδρομένα αεροσκάφη ή ε, οχήματα άνευ οδηγού. Χρειαζόμαστε για αυτά πρόσβαση ε, στο νέφος, αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή στάση. Ο χειρισμός των δεδομένων, όπως είπε η συνάδελφος ε, Σαρτζεντίνη, γίνεται με τον σωστό τρόπο, γίνεται με τον σωστό τρόπο δηλαδή η ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Και αυτό σημαίνει ανωνυμοποίηση. Να μην μπορεί κανείς να επανέλθει στα αρχικά στοιχεία. Γι' αυτό η ανωνυμοποίηση και η ψεύδοανωνυμοποίηση είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα η ψεύδοανωνυμοποίηση στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, παίζει μεγάλο ρόλο. Και παίζει ρόλο να μπορεί να επανέλθει κανείς στα αρχικά στοιχεία για να μπορέσει ακριβώς να του δώσει συμβουλές για την καλύτερη θεραπεία του. Και η αποθήκευση αυτών των δεδομένων δεν είναι τόσο επικίνδυνη. Το θέμα είναι ποιος θα έχει πρόσβαση κατόπιν σε αυτά τα δεδομένα. Θα πρέπει δηλαδή ο τρόπος ε, επαναφοράς στα αρχικά στοιχεία να γίνεται με σωστό τρόπο. Πρέπει να υπάρχει κάποια αρχή που να τα διαχειρίζεται, για παράδειγμα. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο δημιουργικοί όσον αφορά το χειρισμό των στοιχείων και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους. Γιατί αλλιώς πάντα θα είμαστε ουραγοί, θα τρέχουμε από πίσω, τελευταίοι και κατεδρομένοι. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη πρόσβαση. Αν υπάρχουν άλλα μοντέλα πέραν της ε, ψεύδο και άνωνυμοποίησης, ωραία, είμαστε ανοιχτοί. Αλλά χρειαζόμαστε να υπάρχει κάποια ε, πρωτότυπη αντιμετώπιση, ούτω ώστε στοιχεία που αφορούν τα άτομα να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με κάποιες μορφές. Και βέβαια να υπάρχει προστασία μέσω ψεύδο ή και ανωνυμοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να απαντήσει η Κομισιόν σε κάποια Σαλτσεντίνη, που είπε η κυρία Σαρτζεντίνη, αλλά θα ήθελα να απαντήσει στο θέμα του που βρίσκεται αυτό το θέμα του ευρωπαϊκού νέφους του επιστημονικού γιατί βεβαίω η Ήτρε παίζει εδώ τον πρώτο ρόλο και ακούστε τη συζήτηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα από την πτυχή της ιδιωτικότητας για να δούμε πού βρισκόμαστε από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι την Κομισιόν μπορούν να σχολιάσουν αυτή τη στιγμή. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Καλωσορίζουμε τη δουλειά της Επιτροπής σας ε, και την... το σχέδιο έκθεσης για την Επιτροπή Ήτρε. Όσον αφορά την δουλειά που κάνει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν για την ε, δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ανοιχτού Επιστημονικού Νέφους, να πούμε πως η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει μια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για να αξιολογήσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό αυτό επιστημονικό νέφος και να ληφθούν υπόψη όλα τα ζητήματα ιδιωτικότητας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, θα τα δούμε αυτά στο πλαίσιο νέας νομοθεσίας που θα κατατεθεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί δεδομένων. Ε, θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, διαβουλεύσεις και να λάβουμε υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων που επηρεάζονται από την πρωτοβουλία αυτή. Σε σχέση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όλοι βεβαίως ε, είμαστε υπέρ των απόψεων που αναφέρονται στην έκθεση και θεωρούμε ότι μια εναρμονισμένη προσέγγιση στην εφαρμογή του κανονισμού θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε ένα ευρωπαϊκό επιστημονικό νέφος ε, το οποίο θα επιτρέψει την συνεργασία της ε, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας ενώ θα παρέχει διασφαλίσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω κάτι που ανέφερε η Judith Sargentini. Όταν ε, συζητήσαμε την αρχική ιδέα αυτού του νεφούς, είχαμε κάποιες συστάσεις ε, στο τέλος προηγούμενης εντολής και ένα από τα επίμαχα ζητήματα ήταν ότι θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα και ίσως οι συνάδελφοι θυμούνται τις αντιδράσεις ότι προσπαθούσαμε δηλαδή να έχουμε μπει μια αρμονισμένη προσέγγιση που θα ήταν κάποιο είδους φραγμός για ένα νέφος που ουσιαστικά θα ήταν εντός αμερικανικής δικαιοδοσίας αλλά παγκόσμιο και χαίρομαι που άκουσα σήμερα την Adel Γκρίσμπεκ, παραδείγματο χάρη, να λέει και να εκφράζει ολόκληρη την Επιτροπή, νομίζω, από ό,τι άκουσα, ότι έχουμε προχωρήσει πέρα από αυτά τα κλισέ των φραγμών και των τείχων. Τώρα βρισκόμαστε στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Χρειαζόμαστε κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας για αυτό το ανοιχτό επιστημονικό νέφος. Είναι λοιπόν σύντομη η γνωμοδότηση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί η Επιτροπή ΛΥΒΕ πρέπει να εμπλακεί σε αυτά τα θέματα ανωνυμοποιημένων δεδομένων και τη ιδιωτικότητα και να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Νομίζω πως υπάρχει αρκετή εμπειρία σε αυτή την Επιτροπή από την ε, έρευνα και για τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπόνη για να κινηθούμε γρήγορα και να σταματήσει αυτό το κλισέ το ότι χτίζουμε έναν τείχο απέναντι στην Αμερικανική κυριαρχία και ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό νεύος. Υπάρχει χώρος και για εμάς και λόγω του διαδικτύου των πραγμάτων. Και πρέπει γρήγορα λοιπόν να υπάρξει αυτή η εμπειρογνωμοσύνη και βεβαίως ε, έχουμε τα ζητήματα ε, ιδιωτικής ζωής και το νέο κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και είμαι σίγουρος πως θα προσθέσουν συνάλφοι και κάποιες τροπολογίες η Επιτροπή μας. Πολύ σημαντική λοιπόν η συζήτηση και ελπίζω ναι. πως θα παραμείνει και η κληρονομιά εκείνης της εποχής γιατί το είχαμε απορρίψει στις ε, συστάσεις, αλλά είναι στην σύσταση, αλλά είναι κάτι το σημαντικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τον λόγο είχε ο κύριος Μπόνη. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Νομίζω πως έχουμε λίγο χρόνο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο επικοδομητικά χάρη στην συνεργασία μας Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τις ε, συστάσεις μας, το μήνυμα μας από αυτή την πρωτοβουλία και βεβαίως ε, αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων που σχετίζονται με θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία ιδιωτική ζωής και ασφάλεια και είχαμε και τον ε, γενικό κανονισμό και ακριβώς ε, η ακριβής ε, ερμηνεία και κατανόηση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και η ανωνυμοποίηση και η ψευδονυμοποίηση. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για τον νέφος και την θέση του νέφους όταν κοιτάμε τις ψηφιακές εξελίξεις και δεν μιλάμε για τον νέφος το οποίο θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Μιλάμε για έναν έφος το οποίο θα μας επιτρέψει να μοιραζόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα Δηλαδή και τα προσωπικά δεδομένα θα υφίστανται κάποια επεξεργασία. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Μιλάμε για το πώς οι επιστήμονες θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ακριβώ λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασία των Δεδομένων. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και θα πρέπει νομίζω να εκφράσουμε ε, και να περιγράψουμε κάποιες ε, επιπρόσθετες ε, δικλείδες ασφαλείας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία καθορίσατε τον ρόλο μας. Νομίζω πως κάποια πράγματα μάθαμε σήμερα για την ανωνυμοποίηση και την ψευδονυμοποίηση. Περνάμε τώρα στο σημείο 13, την Frontex, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Έχουμε εδώ πέρα τον εκτελεστικό διευθυντή, τον κύριο Φαμπρίς Λετζέρη που έρχεται αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσει όλη μια εισαγωγή λοιπόν. Πρόκειται για παρουσίαση της εφαρμογής του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λετζέρη. Όπως ξέρετε, ο νέος κανονισμός έτεθεν της στις 6 Οκτωβρίου. Έκτοτε ο κύριος Λετζέρη, όπως ξέρετε, Ήδη είχε έρθει σε μια ακρόαση για την Σέγγεν στις 12 Οκτωβρίου και μίλησε για τις αξιολογήσεις ευπάθειας που θα κάνει η υπηρεσία στο μέλλον και τώρα θα μας ενημερώσει για την εφαρμογή του νέου κανονισμού και το σχέδιο πολιετούς προγράμματος. Σύμφωνα με τον κανονισμό άρθρο 64.1 η υπηρεσία θα εγκρίνει ένα έγγραφο προγραμματισμού που θα περιέχει το πολιετές πρόγραμμα για το επόμενο έτος μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της Κομισιόν όσον αφορά τον πολιετή προγραμματισμό, αφού ε, διαβουλευτεί με το Κοινοβούλιο. Για αυτά λοιπόν και για κάποια άλλα οπωσδήποτε που θα ρωτήσουν οι συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και είμαι σίγουρος πως οι συνάδελφοι έχουν κάποιες ερωτήσεις για την υπηρεσία. Θα δώσω λοιπόν στον κύριο Λετζέρη 15 λεπτά να κάνει μια παρουσίαση και μετά θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Λοιπόν, κύριε Λετζέρη, έχετε τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω με μια επισκόπηση για το έγγραφο του πολιτικού σχεδιασμού της Frontex που καλύπτει την περίοδο από το 2017 έως το 2019. Όπως θα θυμάστε, ένα τέτοιο έγγραφο είναι το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό έγγραφο του οργανισμού μας, όπως έχουν όλοι οι οργανισμοί ένα αντίστοιχο. Είναι ένα έγγραφο πολυσέλιδο. Θα προσπαθήσω όμως να πάω στα σημαντικότερα απευθείας. Πώς έχουν τα πράγματα ε, υπολογίζουμε ήδη τι θα συμβαίνει το 2017, αλλά το έγγραφο αυτό θα είναι ένα έγγραφο εν εξελίξη. Θα αναθεωρείται διαρκώ και του επόμενου μήνε και τον επόμενο χρόνο, διότι καλύπτει το διάστημα στο 2019. Βεβαίω, ευχαρίστω θα ξανάρθουμε στο Κοινοβούλιο για να, για να εξηγήσουμε τι θα γίνει με τι μελλοντικέ εξελίξει την ερχόμενη χρονιά. Πρώτον, να εξηγήσω ότι υπάρχουν τέσσερις πολίτες στόχοι οι οποίοι απαριθμώνται. Θα προσπαθήσω να τους εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος που ονομάζεται ευαισθητοποίηση. Η ευαισθητοποίηση σημαίνει ότι ο στόχος του οργανισμού είναι να καταγράφει την κατάσταση της κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης βάσει των μυστικών πληροφοριών που έχουμε και των ε, ε, δεδομένων σε σχέση με τις απειλές για τα, σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν για την ιστορική ασφάλεια της Ένωσης στην περιοχή, στον χώρο ελεύθερης πληροφορίας. Εδώ να τονίσω ότι έχουμε κάποιες συγκεκριμένε δράσεις οι οποίες ε, έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες, έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση του εγκλήματος, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την πρόληψη των τρομοκρατικών δράσεων ε, και στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει ακριβώς ο στόχος της ευαισθητοποίησης όπως είπα. Υπάρχει και αυτός της απόκρισης. Η απόκριση είναι στόχος που έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να διαρματίσουμε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής αντίληψης για την ε, εσωτερική, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ιδίως για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Εδώ οι συγκεκριμένε δράσει μπορεί να έχουν να κάνουν με καταστάσει ε, κατεπίγουσες και την ε, υλική στήριξη των κρατών μελών. Υπάρχει και άλλο ένα στόχο, ο οποίο ονομάζεται ανάπτυξη. Αυτός σχετίζεται με την ανάγκη να αναπτυχθούν καλύτερες πρακτικές, τεχνικός, τεχνική στήριξη, εναρμονισμένα πρότυπα και εναρμονισμένες πρακτικές συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης δηλαδή και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων των κρατών μελών, δηλαδή τη συνεργασία των ομάδων των δυνάμεων δίωξης που προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα. Ο τελευταίο στόχο είναι οι επιδόσει. Ο στόχο είναι να πετύχουμε αποτελέσματα βάσει τη νέα μα του νόμου που άρχισε να ισχύει από τον Οκτώβριο και αυτό έχει να κάνει και με το σεβασμό και την πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διεξαγωγή των ε, αρμοδιοτήτων μα των αποστολών στα εξωτερικά σύνορα. Υπάρχει και μια ε, οικονομική διάσταση, διότι οι επιδόσει εδώ έχουν να κάνουν και με την καλύτερη και πλέον χρηστή διαχείριση των πόρων μα, ώστε να μην υπάρχει υπερβολικό κόστο. Και έτσι όπω μπορεί να εγκρίνεται από τι ευρωπαϊκέ δημοσιονομικέ αρχέ. Αυτά για να εξηγήσω ποιοι είναι οι τέσσερις στόχοι για το διάστημα αυτό, για τον πολιετή σχεδιασμό μας. Τώρα οι στρατηγικοί στόχοι. Έξι στρατηγικές κατευθύνσεις. Στο έγγραφο θα βρείτε ίσως και άλλους όρους να χρησιμοποιούνται, όπως στρατηγική, περιοχές στρατηγικής δράσης. Ξέρω ότι ενός τέτοιου είδους έγγραφο είναι κάπως περίπλοκο λίγο δυσνόητο. Είναι και η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο έρχεται αντιμέτωπο με ένα τέτοιο έγγραφο από τη Frontex, αλλά πραγματικά θα το βελτιώσουμε. Θα το βελτιώσουμε και θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε κατά την ε, εκτέλεση της νέας μας θητείας το περιεχόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε σχεδιασμό του προπολογισμού βάσει των δραστηριοτήτων. Αυτό είναι μια πρώτη έννοια, την οποία δεν θα αναπτύξω εδώ στην παρουσίασή μου, αλλά αν υπάρξουν ερωτήσει, ευχαριστώ να τι απαντήσω. Ερωτήσει οικονομικού περιεχομένου. Πάντω, οι στρατηγικέ κατευθύνσει ω προ το περιεχόμενο είναι οι εξή. Η πρώτη. Η δημιουργία και η ενίσχυση τη τεχνική συνεργασία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Εδώ θα εφαρμόσουμε βάσει της νέας μας θητείας όλα αυτά που μας έχουν ανατεθεί. Με επιχειρήσεις και ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Κάτι που έχει ετοιμάσει ο οργανισμός μαζί με τα κράτη-μέλη. Τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και την δυνατότητα ε, να τα ξανασυζητήσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θα την έχουμε μάλλον και στο μέλλον, αν το επιθυμήσετε εσείς. Θα ήθελα επίσης να τονίσω σε αυτόν τον τίτλο ακριβώς και τις ε, μελέτες για τα ευάλωτα σημεία και την ανάγκη στήριξης των κρατών μελών. Η μελέτη ευάλωτων σημείων είναι ένα νέο στοιχείο που αναπτύσσει ο οργανισμός μας και θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Να τονίσω ότι χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη συνεργασία με, άλλους, ε, με άλλες διοκτικές δυνάμεις όπως την αστυνομία, τελωνιακά, ακτοφυλακές. Ε, έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας όπως είπα, και για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα συμπεριλαμβανομένης τη τρομοκρατίας, Θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο ακριβώς της ολοκληρωμένη διαχείρισης των σύνορων. Να μην το περιορίσουμε στην μετανάστευση. Δεύτερη στρατηγική κατεύθυνση, η ενδυνάμωση της θαλάσσιας διάστασης του οργανισμού. Αυτό είναι ταυτόχρονα συνέπεια και συνιστόσα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των σύνορων, και εδώ, όταν θέλουμε να ε, οργανώσουμε τη συνεργασία μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με άλλους φορείς εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω χάρη με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Θαλάσσια Ασφάλεια, τον Οργανισμό για, την, για τον Έλεγχο των Αλλιευμάτων τα θαλάσσια τελωνία, τον ε, φορέα για, την, ε, για τον τηλεφωνικό έλεγχο σε θαλάσσιες οδούς, όλα αυτά είναι θέματα που εντάσσονται εδώ. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα ε, άπτεται και της ε, διάσωση και θα έχουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να συνεργαζόμαστε καλύτερα είτε στο πλαίσιο των κοινών μας επιχειρήσεων όπως του Τρίτονα και του Ποσειδώνα κάτι που ήδη έχουμε κάνει, είτε να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες όπου χρειάζεται. Τρίτη στρατηγική κατεύθυνση. Διαχείριση της μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα. Θα υπάρχουν ειδικέ ομάδες στήριξης για τη μετανάστευση, αυτή είναι μια νέα έννοια, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών hot spot, κέντρων υποδοχής, που θα είναι καλύτερα οργανωμένα, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στο, ε, στην έμαστε εντολή. Τέταρτη στρατηγική κατεύθυνση, επιστροφές. Εδώ ο οργανισμός θα εξετάζει τις ομάδες που είναι υποχρεωτικές βάσει του νεοκανονισμού, όπως αυτές της ε, συνοδείας, της ε, παροχής στήριξης και επίσης θα παρέχεται και αρρωγή στα κρατημέλη για τον εντοπισμό υπηκών τρίτων χωρών και για να αναπτύξουμε βαθμιδών καλύτερες και πιο συντονισμένες προσεγγίσεις μεταξύ των διαφορών κρατών μελών αλλά και των διαφορών φορέων και υπηρεσιών εντός των ιδίων των κρατών μελών με στόχο να έχουμε πιο ολοκληρωμένη, πιο ενοποιημένη διαχείριση των επιστροφών. Εδώ θα συμπεριλαμβάνεται και διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι που αντικατοπτρίζεται συνολικά στις δραστηριότητες του οργανισμού. Πέμπτη στρατηγική κατεύθυνση. Συνεργασία με τρίτες χώρες όπως ορίζει η νέα εντολή που έχει ανατεθεί στον οργανισμό μας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τους εξωματικούς συνδέσμους και την αποστολή τους σε τρίτες χώρες, κάτι που ξεκίνησε ήδη φέτος, πριν την έναρξη υλοποίηση της νέας εντολής. Έχουμε έναν αξιωματικό σύνδεσμο στην ε, Τουρκία, αλλά τώρα αυτό θα επεκταθεί ω μέτρο. Η στρατηγική τώρα σχεδιάζεται εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ε, για τις τρίτες χώρες ενώ και θα προβλέπεται η δυνατότητα να αποσταλούν, να οργανωθούν μάλλον κοινέ επιχειρήσει με τρίτε χώρε. Θα ληφθεί και αυτό υπόψη και θα ενταχθεί σε αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση. Έκτη και τελευταία στρατηγική κατεύθυνση που μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο αυτό είναι η ενδυνάμωση και επέκταση των ε, δραστηριοτήτων οικονομικής ε, διαχείριση του οργανισμού, για τον τεχνικό εξοπλισμό και του ανθρώπινου πόρου, όπω διατίθενται από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στη διαχείριση αυτών των πόρων. Η αγορά του τεχνικού εξοπλισμού του ίδιου του οργανισμού εντάσσεται εδώ και υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με την κατάρτιση και την εκπαίδευση, τις σχετικές πολιτικές του οργανισμού και την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μέλη τα οποία είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα και έχουν τι κατάλληλε επιδόσει και στη συνοριοφυλακή και στην ακτοφυλακή. Αυτέ ήταν οι βασικέ θετικέ κατευθύνσει. Τώρα μια επισκόπηση των προσφατότερων μέτρων που έχουν ε, ληφθεί για την υλοποίηση, την εκτέλεση της εντολής, η οποία αρχίζει να ισχύει από τις 6, έχει αρχίσει να ισχύει από τις 6 Οκτωβρίου, στις επιστροφές. Έχουμε αναπτύξει και άρχισε να λειτουργεί ε, ένα σύστημα αιτήσεων για τις επιστροφές ε, στα κρατημέλη, ένα σύστημα ηλεκτρονικό που έχει οργανώσει η Επιτροπή με τα κρατημέλη. Εκεί τα κρατη μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους στο σκέλος των επιστροφών. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό προσφυγών, έχουμε ανεβάσει στον ιστότοπο του οργανισμού ένα έντυπο για τις προσφυγές, για όσους θα θέλαν να υποβάλουν προσφυγή. Όλα τα σχετικά έγγραφα και κανόνες που διέπουν το μηχανισμό προσφυγών είναι στον ιστότοπο. Αυτό που λείπει είναι το δίκτυο των σημείων επαφής των κρατών μελών, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και ανεξάρτητα από τους φορείς ακτοφυλακής, δηλαδή τα κρατημέλη θα πρέπει να κάνουμε και κάτι εδώ, ώστε και ο αξιωματικό για τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατών μελών του οργανισμού να μπορεί να έρθει σε επαφή με τι εθνικέ ε, αρχέ. Και επίση. Υπάρχει σχετική εκπαίδευση για να καλυφθεί και η γλωσσική διάσταση. Τώρα για την ε, ακτοφυλακή. Ήδη διαπραγματευόμαστε το σύστημα εργασία που θα έχουμε σε συνδυασμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για Θαλάσσια Ασφάλεια και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αλίας. Έχουν προχωρήσει συζητήσει. συζητήσεις. Υπάρχει περισσότερη επιχειρησιακή συνεργασία με ένα πιλωτικό πρόγραμμα του οργανισμού, για... του οργανισμού που παρακολουθεί την παράνομη και παράτυπη αλία Εδώ λοιπόν η παράνομη αλία είναι ένα από τα πράγματα που αναφέρει το έγγραφο και είναι ένα τομέα που δεν μπορούσαμε να δραστηριοποιηθούμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί προ το κόστο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και την πρώτη πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ακτοφυλακών. Ένα καινούριο δίκτυο που αρχές δίωξης με αρμοδιότητες στη θάλασσα συνεργάζονται πλέον μεταξύ τους. Για τη μεθοδολογία των μελετών ευάλωτων σημείων αγκρίθηκε τον Οκτώβριο το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική μεθοδολογία και είναι εν εξελίξει συζητήσει με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Την ερχόμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει πρόταση από τον εκτελεστικό διευθυντή με περισσότερε λεπτομέρειε για τους στόχους της επόμενης χρονία. Από τα κάτι μέλη αυτό που αναμένεται είναι να διορίσουν εκπροσώπους στο δίκτυο για τις μελέτες ευάλωτων σημείων. Οι ομάδε. και ανθρώπινοι πόροι του θα ε, οργανωθούν εγκαίρω. Ήδη η σύνθεση κάποιων από αυτέ εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, προϋπόθεση πριν οργανωθούν κοινέ επιχειρήσεις με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε τρίτες χώρες, είναι η ολοκλήρωση του ε, προτύπου συμφωνίας που θα ισχύσει για τις περιπτώσεις αυτές, αυτό να το κάνει η Επιτροπή σε συνεργασία με τον οργανισμό και να είναι σαφές ότι από την οπτική γωνία του οργανισμού και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι και από την οπτική γωνία των κρατών μελών αυτό που προέχει είναι να υπάρχει νομική προστασία των αξιωματικών μα που είναι σε τρίτες χώρε αλλά και των ε, περιουσιακών μα στοιχείων. Να μην χρειαστεί επίση να πληρώσουμε τασμού, ξέρω εγώ, βασικό στοιχείο. Αλλά πρέπει να καλύπτεται στην ε, συμφωνία μοντέλο που θα ισχύσει. Για το Διοικητικό Συμβούλιο ε, να πω ότι ενέκρινε την προτινόμενη στρατηγική ω προ τη γεωγραφική κατανομή των αξιωματικών συνδέσμων που θα αποσταλούν στον Ήγηρα στην περιοχή των Βαλκανίων και το επόμενο κύμα είναι άλλες χώρες της Βορείου και της Δυτικής Αφρικής, του κέρατος της Αφρικής, και σε άλλες περιοχές. για τα επιχειρησιακά. Σύντομα θα προταθεί η επιχειρησιακή στρατηγική και να μιλήσω και για τις προσλήψεις και το πώς έχουν εκεί τα πράγματα. Ξέρω ότι συζητιέται αυτό στο Κοινοβούλιο για το front loading, την εμπροστοβαρή προσέγγιση. Αυτό σχετίζεται με τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου, αλλά η ιδέα ήταν ε, να προβλέψουμε προκαταβολικά 50 θέσεις και να τις πληρώσουμε από τις 250 που πρέπει από την Επιτροπή για το 2017. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προσλήψεις και έχουμε εντοπίσει τους κατάλληλους υποψηφίου. Τους προσφέραμε λοιπόν τα σχετικά πόστα. Σε ό,τι αφορά, και αυτό θα είναι το τελευταίο μου παράδειγμα, διότι μάλλον μακρηγόρησα, σε ό,τι διαφάνεια και το, υπολο, το, τη λογοδοσία, το έχω ξαναπεί στην Επιτροπή Λίμπα. Περισσότεροι πόροι και αρμοδιότητε για τον οργανισμό μα σημαίνουν και περισσότερη λογοδοσία. Έχουμε βελτιώσει αυτό το σκέλο. Πρόσβαση στα έγγραφα λόγου χάρη. Υπηρεσία διαφάνεια εντό του οργανισμού για να αποκρινόμαστε καλύτερα στα σχετικά αιτήματα για πρόσβαση στα έγγραφα. Τη δημόσια πρόσβαση εννοώ. Την πρόσβαση του κοινού. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων ως προς την εκτέλεση της νέας εντολής. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις εφόσον υπάρξουν. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Λετζέρη. Ε, θέλουμε να μας μιλήσετε για την εφαρμογή του κανονισμού κυρίως, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι μπορεί να θέσουν και μερικά ευρύτερα θέματα που σχετίζονται με τον οργανισμό σας. Ελπίζω να έχετε κάθε διάθεση να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο για να θέσουν ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μιλήσουν πρώτοι και συντόμως παρακαλώ οι σκιώδεις για τον κανονισμό και μετά θα δώσω το λόγο και σε άλλους. Συνάδελφοι σας παρακαλώ, δύο λεπτά ο καθένας για να μπορέσουμε να λάβουμε και απαντήσεις ουσιώδεις. Γιατί ξέρω ότι έχουν τεθεί μερικά πολύ σημαντικά θέματα πρόσφατα για τον οργανισμό αυτό και τη λειτουργία του. ισχυώδης λοιπόν για τον κανονισμό. Ναταλή Κρισμάν. Κρισμπέκ, συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λεζερή για την παρουσία σας. Πάντα πολύ σαφής. Θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι ιδιαίτερα ε, για τις ε, νέες αρμοδιότητες και αποστολές αυτού του νέου οργανισμού, γιατί θεωρώ ότι είναι νέος. Ακόμη και αν ε, η κοινή γνώμη δεν καταλαβαίνει πάντα ότι είναι ένας νέος οργανισμός με νέες δυνατότητες. Αντίθετα, οι συμπολίτε μας, πολλοί από αυτούς τουλάχιστον, θεωρούν ότι αυτό το νέο σύστημα θα τα λύσει όλα τα προβλήματα. Εγώ από πλευρά μου, όταν τους εξηγώ τον τρόπο λειτουργίας και ότι είμαστε σε φάση εκκίνησης ε, του νέου οργανισμού, τους εξηγώ τη σημασία και τις διαστάσεις της πρόκλησης, αλλά βεβαίως προσπαθώ αναλυτικά να τους εξηγήσω ότι δεν θα τα λύσει και όλα. Δεν θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσχέρειες στα εξωτερικά μας σύνορα. Ίσως να μας επιτρέψει όμως ε, να εδραιώσουμε το σύστημα Σέγγεν και την ελεύθερη κυκλοφορία. Δύο-τρεις σύντομες ερωτήσεις. Και είπα ήδη ότι χαίρομαι για τη λειτουργία αυτής ε, της ε, νέας μορφής αντιμετώπισης, αλλά ίσως να θεωρήσετε παρόλα αυτά ότι είναι λίγο δυσάρεστες οι ερωτήσεις μου. Αναφερθήκατε στις επιστροφές. Πολλοί εκφράσαμε ανησυχίες για αυτές τις, ε, τις δραστηριότητες που διεξάγονται στα σύνορα. Δηλαδή, ορισμένα άτομα επιστρέφονται απευθείας στα σύνορα. Γιατί νομίζω ότι είναι ασαφής ε, η κατάσταση εκεί, μπορεί να διατρέχουν κινδύνους και μπορεί να εφίστανται κακοποίησεις. Υπάρχει κακοποίηση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θα μου πείτε βέβαια όχι. Αλλά θέλω να πω υπάρχουν άτομα που αποθούνται χωρίς να έχουν δυνατότητα να υποβάλουν το αίτημα ασύλου σε κάποιο κράτος μέλος. Ισχύει αυτή η αντίληψη που κυκλοφορεί. Δεύτερη ερώτηση, επίσης δυσχερής. Υπήρξαν διάφορα επεισόδια που έχουν να κάνουν με τη χρήση όπλων από τους ακτοφύλακες στα πλαίσια της λειτουργίας. Και ιδιαίτερα ακούστηκε ότι πυροβόλησαν και ορισμένα σκάφη με πρόσφυγες. Φυσικά τα σκάφη αυτά τα οδηγούν διακινητές, οι οποίοι είναι βέβαια άθλοι. Θέλω να μας δώσετε εξηγήσεις. Και τρίτη ερώτηση, που ξέρω ότι και αυτή είναι δυσχερής, τι γίνεται με την κατάσταση ακριβώς ε, ανοιχτά των τουρκικών ακτών, που είναι τα σύνορά μας. Ευχαριστώ. Η Σκά η δεύτερη σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Ριζερή που ήρθατε και μας εξηγήσατε την εφαρμογή της εντολή της εντολής σας για το μηχανισμό προσφυγών ή παραπώνων. Είπατε ότι υπάρχει δυνατότητα στο ίντερνετ. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν σημεία επαφή με τα κράτη-μέλη. Δεν σας δίνουν. Δεν έχουν κάποιον που θα είναι κατάλληλο γι' αυτό. Επίσης, θεωρώ ότι θα ήταν καλό αυτός ο μηχανισμός ε, να είναι σε ένα πιο εμφανέ σημείο του, της ιστοσελίδας σας και δεν μπορεί κανείς ούτε επιγραμμικά να τη συμπληρώσει. Καλύτερα θα ήταν λοιπόν να μην είναι μόνο για τα μάτια. Είναι πολύ δύσκολο να τη βρει κανείς τώρα αυτή την... Τη, να βρει κανείς αυτό το έντυπο. έντυπο. Και επίσης, ο αρμόδιος ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προσφυγές. Το Κοινοβούλιο είπε ότι πρέπει να έχει επαρκές, ε, επαρκές δυνατότητες, επαρκές προσωπικό πόρους. Πού θα είναι αυτό το, πού θα είναι αυτή η μονάδα για αυτήν την ε, ομάδα για, τα, για την συνοριοφυλακή. Τι γίνεται ακριβώ με αυτή την ομάδα. Υπάρχουν κράτη-μέλη που να έχουν δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχουν με ακριβή αριθμό ή με κάποιο αριθμό συνοριοφυλάκων και για τις τρίτες χώρες. Με ποιες τρίτες χώρες ε, σκοπεύετε να συνεργαστείτε. Νιζέρ, Βαλκάνια, Βόρεια και Δυτική Αφρική, αυτές που ήδη αναφέρατε. Και ποια είναι η τελευταία χώρα που είπατε. Μετά από τη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική δεν το ακούσαμε. Και τι ακριβώ θέλετε να κάνετε με αυτέ τι χώρε. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις επαναπροώθησης από την Ελλάδα, όπου γίνεται μελέτη, ε, έρευνα από τις ελληνικές αρχές, που έγιναν με τα μέσα του Frontex. Δηλαδή με ένα αεροπλάνο το οποίο ε, μίστοσε η Frontex. Ε, τώρα ξέρετε, αν γίνεται με μίσθωση της Frontex, με προσωπικό τη Frontex, φαίνεται να τα κάνει, σαν να τα κάνει όλα η Frontex. Δεν θα πρέπει κάτι να αλλάξει για να μην υπάρχει αυτή η εντύπωση. Και επίση οργανώσατε μια συνδιάσκεψη για την ακτοφυλακή πρόσφατα, πριν δύο μέρε. Και προσκαλέσατε για την Αυστραλία. Τι θέλετε να μάθετε από την Αυστραλία και από την στο ακτοφυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Αρκετές ερωτήσεις, ελπίζω να τις σημειώσατε, λέει ο κύριος ε, Μωράς. Και σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να ακούσω και τις απαντήσεις. Επειδή πολλοί θα κάνουν παρόμοιες ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων. Λοιπόν τώρα, με τη σειρά ε, αυστηρά που ζητήθηκε ο λόγος. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κλοντ. Κύριε Λεζερή, καλώ ήρθατε. Πάντα είναι ευχαρίστηση να συζητάμε και γιατί είναι πάντα σαφής αλλά και σωστά δομημένη η παρουσίασή σας. Τρει ερωτήσει. Δεν θέλω να προκαλέσω σύγχυση μεταξύ ανομίων πραγμάτων, αλλά διάβασα μια έκθεση στην εφημερίδα Le Monde πριν από μερικέ μέρε. Μια πολυσέλιδη έκθεση και έλεγε ότι μεταξύ των τρομοκρατών που ε, έκαναν ε, τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι και, τη, και στις Βρυξέλλες. Οι περισσότεροι ήταν μαχητές στη Συρία και επέστρεψαν παράνομα στις χώρες μας. Δεν κάνω, δεν κάνω καμία εξομοίωση μεταξύ μεταναστών και τρομοκρατών και αυτά τα λέει μια εφημερίδα που δεν θεωρείται ιδιαίτερα δεξιά. Και βεβαίως εκτιμώ την εργασία του συντονιστή για τα θέματα αυτά της Europol, αλλά είναι χιλιάδες μαχητές που υπάρχει κίνδυνος να επανέλθουν στην Ευρώπη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και το Ιράκ. Θεωρείτε ότι έχουμε επαρκές πλαίσιο ούτως ώστε στα σύνορα να παίξουμε ουσιώδη ρόλο για να επιλέξουμε ε, αυτούς που θα μας δημιουργήσουν προβλήματα για να τους διαχωρίσουμε από τους άλλους. Δεύτερον, κάτι που έχει να κάνει με την ε, σημερινή συγκυρία ο Βέλγος υφυπουργό για τη μετανάστευση που είναι κάπως ιδιαίτερος ανακοίνωσε δημόσια ότι θα ανακαλέσει όλους ε, τους Βέλγους υπαλλήλου που έχουν ε, αποσπαστεί στην Ελλάδα γιατί μας είπε, έχει προφορίες ότι η ασφάλειά τους δεν, έχουν, ε, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται βεβαία ότι επιτέθηκαν ορισμένοι μετανάστες ε, σε κτίρια όπου εργάζονται αυτοί και ότι τους απειλούν κάποιοι καθημερινά. Είναι αξιόπιστα αυτά τα στοιχεία, τέτοιου τύπου γεγονότα έλαμα χώρα. Και αν ναι, τι ε, πορίσματα εξάγεται. Ευχαριστώ πολύ, για Πρόεδρος. Η Κριστίν Ντελάνη. Ευχαριστώ, κύριε Λεντζέρη για την παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, δύο σημεία συγκεκριμένα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των συνδροφυλάκων και αποφυλάκων, όπου θα ισχύσουν διατάξεις του νέου κανονισμού. Οι δραστηριότητε, οι ειδικέ δραστηριότητε κατάρτιση που έχουν να κάνουμε παιδιά και άλλα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση, άρθρο 36 έχουν ήδη σχεδιαστεί αυτά. Και δεύτερον, ήθελα να επιμένουμε λιγάκι στι συμφωνίε συνεργασία με τρίτε χώρε, στι οποίε πολύ συχνά στέκομαι και σα θέτω ερωτήσει. Μεταξύ των εγγράφων για την συνεδρίαση σήμερα, λάβαμε και την συμφωνία που υπογράφηκε με το Κωσυφοπαίδιο στι 25 Μαου του 2016. Ε, το στοιχείο του κειμένου αυτό έχουν ήδη διατεθεί στο διαδίκτυο και μπορεί να τα δει κανεί, όμω το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται συστηματικά για τι ε, συμφωνίε συνεργασία με 18 χώρε. Πώ να το εξηγήσουμε αυτό, μπορείτε να μα δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασία με τρίτε χώρε στα πλαίσια αυτών των ε, συμφωνιών, ε, ιδίω μετά τη συμφωνία που συνήφθη με την Τουρκία, για να αναφέρω μόνο αυτή. Σε ό,τι αφορά τον πολιετή προγραμματισμό του οργανισμού για την περίοδο 2017-2019, ε, αναφέρεται ότι οι περισσότερε ε, συμφωνίε συνεργασία που ισχύουν θα πρέπει να ε, αναθεωρηθούν βάσει του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνεροφυλακή και Ακτοφυλακή και βάσει των κοιτάξεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η διαδικασία αυτή αναθεώρηση των συμφωνιών συνεργασία έχουν αναθεωρηθεί και πώ θα τροποποιηθούν προκειμένου να συνάδουν με τον νέο κανονισμό και την ε, υποχρεω... τον υποχρεωτικό σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο θέλει να τηρείται ενήμερο για την διαδικασία αυτή αναθεώρηση και σύμφωνα με το άρθρο 52 του νέου κανονισμού, ο οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο πριν τη σύναψη συμφωνία συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι θα αποστέλλονται στο Κοινοβούλιο πληροφορίες πριν τη σύναψη συμφωνιών ή για αυτές που τώρα έρχεται με τη Σενεγάλη, την Μαυριτανία, τη, Λιβ... τη Λιβύη, την Αίγυπτο και άλλες χώρες ε, και οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα γνωρίζει γέρο το Κοινοβούλιο τι συμβαίνει στι διαπραγματεύσεις με τρίτε χώρες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λετζέρη για τι πληροφορίε που μας έδωσε. Απλά αναρωτιέμαι, εγώ είμαι τώρα δυόμιση χρόνια εδώ βουλευτή. Ξεκινήσαμε με την επιχείρηση Mare Nostrum, μετά είχαμε την Frontex, ε, τριπλασίασαν τα κονδύλια τους για να αναλάβουν και τις αρμοδιότητες της Mare Nostrum. Τώρα έχουμε νέα Frontex. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω τι γίνεται εντάξει, να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας ε, σύνορα, αλλά η Frontex κατά 98% κάνει έρευνα και διάσωση. Οπότε να ρωτιάμε, η νέα Frontex θα προστατεύσει τα σύνορά μας ή πάλι κατά βάση θα κάνει έρευνα και διάσωση. Άλλη ερώτηση. Στη Σουηδία δεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών πέρσι ο Υπουργός μας είπε ότι η πρόθεση είναι να επιστραφούν τουλάχιστον 80.000. Ε, αναρωτιέμαι λοιπόν, ο, καθώς λέτε πως υπάρχει νέα Frontex, μήπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τα κράτη-μέλη να εκφράσουν ανάγκες που έχουν για βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ε, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε και με αυτό το θέμα, την, ε, τους 80.000 δηλαδή στην Σουηδία. Ένα άλλο θέμα το οποίο διάβασα σήμερα είναι ότι η Ιταλία δέχεται ε, υψηλές πιέσεις ε, ε πέρα από την Ελλάδα μέσω Τουρκίας και διαβάζω ότι η Τουρκία τους η, η Ιταλία τους τελευταίους μήνες έχει αφήξεις ρεκόρ και ε, ακούγαμε πέρσι τα προβλήματα που είχαμε με την έρευνα και διάσωση με επιθετικούς διακινητές ε, που χρησιμοποιούσαν όπλα κτλ. Και αναρωτιέμαι τι θα κάνει η νέα Frontex ε, για αυτό. Γιατί υπάρχουν νέες ροές και από αυτή την πλευρά. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν. Σας ευχαριστώ κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι υπήρχε μια μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για να γνωρίσουμε πως τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών σε ένα βαθμό είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή φυλακή και ακτοφυλακή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ερώτηση για το τι συμβαίνει τώρα στην πράξη. Αντιλαμβάνομαι πως ένα από τα καθήκοντά σας είναι να συλλέγετε δεδομένα, να αναλύετε το τι συμβαίνει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τι κάνετε με αυτές τις πληροφορίες όμως. Γιατί μιλήσατε για το ότι θα ελέγξετε αν υπάρχει αντίκτυπος στην ασφάλεια των συνόρων ε, και την στιγμή ακριβώς που υπάρχει αντίκτυπος στην ασφάλεια των συνόρων μας ίσως να είναι κάπως αργά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με βάση τις αναλύσεις σας για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης και τελικά να καταλήγει αυτό το πράγμα στα σύνορά μας. Αναφέρατε και τη συνεργασία με τις ε, τρίτες χώρες. Σε τρίτες χώρες δεν ε, πάτε για να πολεμήσετε το έγκλημα ή να ενισχύσετε τη δημοκρατία, είναι για να ενισχύσετε τα σύνορα αυτών των χωρών ή κάντε κάτι άλλο εκεί. Οπότε και πάλι το ερώτημά μου είναι με βάση τις αναλύσεις σας δίνετε πληροφορίες σε άλλους κλάδους της Κομισιόν και στα κράτη-μέλη γιατί Όλα αυτά ξεκινάνε, πολλά από αυτά ξεκινάνε σε τρίτες χώρε. Με βάση λοιπόν τι δικέ σα αναλύσει και αναλύσει άλλων υπηρεσιών και εθνικών υπηρεσιών, εγώ νομίζω πω οι προφορίε σα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρο μια στρατηγική για να συνεργαστούμε καλύτερα με τρίτες χώρε για να βελτιωθεί η κατάσταση ή τουλάχιστον να μην επιδεινωθεί καταστάσεις ε, συγκρούσεων, ε, αυταρχικών καθεστώτων, βασανιστήριων και οικονομική κατάσταση ίσως. βοηθούν οι αναλύσεις σας και σε, αυτή, σε αυτόν τον τομέα ή εσείς περιμένετε μέχρι να φτάσει η κατάσταση στα σύνορα και μόνο τότε μπορείτε να αντιδράσετε. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ δόκτωρα Λετζέρη για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις για συγκεκριμένα επεισόδια χρήσης βίας. Το πρώτο, αυτό που αναφέρει και για την παράνομη δίαιη ε, επιστροφή από την Ελλάδα στην Τουρκία με την παρουσία δύο σκαφών της Frontex στις 16 Ιουνίου. Η απάντηση της Frontex ήταν ότι η απόφαση ελήφθη από το Κέντρο Συντονισμού στην Ελλάδα. και βάσει τη ισχύουσα νομοθεσία και μετά από εντελεχή αξιολόγηση τη κατάσταση. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι ποια η ευθύνη της Frontex παρόλα αυτά. Και τι σημαίνει αυτή η εντελεχής ε, εξέταση του θέματος εντελεχή αξιολόγηση. Πώ προχωρήσετε σε αυτή τη βία η επιστροφή, την αναγκαστική επιστροφή. Η δεύτερη παρατηρήσή μου αφορά την καταγγελία της Amnesty International για τη χρήση βίας και βασανισμών σε μια σειρά από κέντρα υποδοχής στην Ιταλία από hot spot στην Ιταλία. Οι αρμόδιες Ιταλικές αρχές τηρούν σιγή ηχθείως από αυτού. Και είναι οι κατεξοχήν αρμόδιες, έτσι. Η ερώτηση είναι, η Frontex προσφέρει αρρωγή στη φάση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες σε αυτή την περίπτωση. Εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη από ό,τι έχω και να μου την πείτε. Τρίτη περίπτωση, η χρήση βίας, χρήση πυροβόλων όπλων επί των σκαφών μεταναστών στην Ελλάδα, όπως καταγγέλει η Intercept τον Αύγουστο φέτος. Ε, σε ένα γράμμα που έλαβα εγώ ως απάντηση είναι ότι δεν υπήρχαν σκάφη της Frontex στην όλη ιστορία. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά η δημοσιογράφος που έκανε την έρευνα, η δημοσιογράφος της Intercept, για να ανέβει στα σκάφη, χρειάστηκε να ζητήσει άδεια τη Frontex. Άρα, σκάφη της Frontex υπήρχαν ή δεν υπήρχαν. Τι έγινε τελικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. And Mr. Kirkos, Ευχαριστώ κύριε Κύρκος. Welcome, Mr. Καλώς ήρθατε κύριε Λεζερή. Πάντα είναι χαρά μας να σας βλέπουμε. Το 2010 υπήρχε μεγάλη είσοδος ε, μεταναστών από την Τουρκία και προσφύγων και η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε μια απόφαση που καταδίκαζε την κυβέρνηση ότι δεν σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αξιοπρέπεια των μεταναστών. Η Frontex είχε 175 άτομα προσωπικό τότε. Και είχε έμεση σχέση με την περίπτωση. Τώρα σε έρθουμε στο σήμερα. Μας είπατε ότι θέλουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Και επίσης ότι θέλετε να αξιολογούμε τα hotspot ε, και ποια έχουν προβλήματα και τι δυνατότητες και δυναμικό έχουν τα κράτη-μέλη και ότι όταν υπάρχει ανάγκη θα υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο. Αλλά τα hotspot μπορεί να δημιουργούν προβλήματα και για τη δυνατότητα χορήγησης ασύλου και επίσης να μην έχουν δυνατότητα να χορηγήσουν τροφή και διαμονή σε όλους. Τι διδάγματα ε, εξήχθησαν από την ελληνική περίπτωση. Έχουμε μηχανισμό για να εντοπίζουμε και να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα αλλά βεβαίως θέλουμε να βοηθήσουμε τη Frontex και είμαστε αισιόδοξοι για τη λειτουργία της αλλά τελικά η αντιμετώπιση που υπήρξε στην Ελλάδα δεν έδωσε αποτελέσματα. Στην Ελλάδα ακόμη ζουν σε πολύ δυσχερείς συνθήκες. Μήνες μετά τον εντοπισμό του προβλήματος δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν έχει επιληθεί. Πώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι, ότι θα έχει αποτελέσματα η λειτουργία της Φράνταξ ε, και δεν θα αρχιοθετούνται ορισμένα θέματα που τίθενται χωρί να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Νάγκη. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που ήρθα μόλι τώρα, ήμουν αλλού. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Σας παρακαλώ, εξηγήστε μου. Τι συμφωνίες χρειάζεστε. Τι συμβάσεις, τι διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ή με διεθνείς οργανισμούς, οργανισμούς ε, των ΗΠΑ Εθνών. Για να υπάρξει πραγματική δράση. Στην άλλη πλευρά της Μεσογείου. Για να αποφύγουμε η να ε, παρεμποδίσουμε την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την δραστηριότητα διακινητών. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, ο για καταπληκτικές ερωτήσεις, για τον κανονισμό. Κύριε Λεζέρη, είστε έμπειρος. Ξέρετε ότι σε αυτή τη συγκυρία ε, είναι πολύ σημαντικό να απαντηθούν πολλά θέματα που έχουν μείνει αναπάντητα. Νομίζω ότι σας αφήσαμε αρκετό χρόνο για να συζητήσετε και να ασχοληθείτε με τα σημαντικά θέματα που τέθηκαν. Σας παρακαλώ με την ησυχία σας, αν θέλετε να απαντήσετε με λεπτομέρειες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που έκαναν ερωτήσεις. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον τους και θα προσπαθήσω να απαντήσω λεπτομερώς θα προσπαθήσω να απαντήσω και στο μετρό δυνατού στην γλώσσα του κάθε βουλευτή. Να μιλήσω και γαλλικά και αγγλικά και... Λοιπόν, για τις ε, επιχειρήσεις επιστροφών, στα σύνορα δηλαδή, pushback, και αν έχουν υπάρξει καταχρήσεις και αν άτομα δεν είχαν δυνατότητα να υπογάλουν αίτηση ασύλου. Νομικά υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέμε η επιστροφή ή η απομάκρυνση. Αυτό γίνεται με βάση την οδηγία 115 του 8, δηλαδή άτομα σε παράτυπη κατάσταση σε μια χώρα της Ένωσης που μετά από την ε, διαδικασία, μετά το τέλος μιας ολόκληρης ε, ε, διοικητικής διαδικασίας επιστρέφονται σε μια τρίτη χώρα. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή που περιγράψατε. Δηλαδή δεν γίνεται είσοδος τους. Με βάση την, ε, τον κώδικα για τα σύνορα του Σέγγεν υπάρχει μια διαδικασία. Όταν ένα ξένος που δεν είναι πολίτης της Ένωσης και που δεν μπορεί να αποφεληθεί από την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη, εάν το άτομο δεν πληρεί τα κριτήρια, δεν έχει βίζα, δεν έχει διαβατήριο, δεν έχει ισχύοντα έγγραφα, εάν δεν πληρεί ορισμένες συνθήκες ιδιαίτερα οικονομικές ή αν προφανώς βεβαίως ε, ε περιέχεται στο σύστημα σέγγεν, στο σύστημα των σεσμασμένων ατόμων, τότε φυσικά ε, μπορεί να το απογορευτεί είσοδος. Εάν ένα άτομο λοιπόν δηλώσει ότι έχει ανάγκη προστασίας, τότε με βάση και την εκπαίδευση που έχουν οι συνοριοφύλακες ή οι ακτοφύλακες, τότε έχει δυνατότητα να του δώσει πρόσβαση και να το στείλει στις αρχές που ασχολούνται με το άσυλο. Ορίστε λοιπόν. Στα πλαίσια των, ε, της δραστηριότητας του Frontex δεν έχω στοιχεία περιπτώσεων όπου συνοριοφύλακές μας να έκαναν κάτι παράτυπο. Έχω ακούσει από ορισμένε ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, έχω λάβει ε, μηνύματα και οποτεδήποτε υπάρξει κάτι τέτοιο αρχίζουμε όσο μπορούμε έρευνες. Σε αυτή τη φάση εξετάζω προσεκτικά ορισμένες ε, καταστάσεις που μπορεί να έχουν προκύψει σε κάποια χερσαία εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω περιπτώσεις στοιχειοθετημένες. Τώρα έγιναν ερωτήσεις για τη χρήση πυροβολών όπλων. Είναι λίγο παράδοξο να απαντήσω γι' αυτό. Να χρειάζεται σήμερα να απαντήσω. Γιατί τα μάθατε χάρη στην πολιτική διαφάνεια της Φράντεξ, την οποία εγώ θέλησα να εισαγάγω. Υπάρχουν περιπτώσεις. Υπήρξαν περιπτώσεις, πολύ άριθμες στην Ελλάδα, ή περιπτώσεις όπου πυροβόλησαν τους συνοροφύλακες, γιατί συνήθως γίνεται ανταλλαγή πυρών. Πυρά και προς τις δύο περιπτώσεις προς τις δύο κατευθύνσεις. Από το καλοκαίρι του 2015 και αργότερα, στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στα όρια των ε, ελληνικών και ε, τουρκικών υδάτων, ε, χωρίων υδάτων, υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα σκάφη μας ήταν πολύ κοντά, χωρίς όμως να έχουν εμπλακεί στις περιπτώσεις ανταλλαγής προφορισμών. Θέλησα να σε ενημερώσω γι' αυτό, όπως ενημερώσαμε και έναν δημοσιογράφο και ο δημοσιογράφος ενώ του δώσαμε πρόσβαση σε έγγραφα, μετά είπε ότι α, είναι έγγραφα που διέρευσαν. Αυτό είναι απόλυτα ψευδές. Του τα δώσαμε τα έγγραφα αυτά. Βέβαια αυτό δημιουργήσε κάποιο ενδιαφέρον, γιατί υπήρξε, υπήρξαν πυροβολισμοί. Οι πυροβολισμοί στην Ελλάδα συνέβησαν με βάση την ελληνική νομοθεσία. Ε, γενικεύοντας λιγάκι για τις επιχειρήσεις της Frontex στο επιχειρησιακό μας σχέδιο υπάρχουν διατάξεις που αφορούν την νόμιμη άμυνα και ο κανονισμός αυτός για την νόμιμη άμυνα δεν είναι ο ίδιος για παράδειγμα μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας μπορούν να υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα αλλά λοιπόν, στα σκάφη και στους ακτοφύλακες που δεν είναι υπήκοοι του κράτους όπου δρούν, δηλαδή οι μη Έλληνες στην Ελλάδα και οι μη Ιταλοί στην Ιταλία, τους συστήνουμε να μην παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί να πυροβολήσει κάποιος. Να μην πυροβολούν δηλαδή εκείνοι. Αλλά φυσικά αν τους πυροβολούν, έχουν δυνατότητα να πυροβολήσουν με βάση και το εθνικό δίκαιο. Όμως κανένα σκάφος της Frontex δεν ενεπλάκησε τέτοιους πυροβολισμούς και από ό,τι καταλαβαίνω από τις εκθέσεις των ερευνών που ζήτησα και μου έδωσαν ελληνικές αρχές δεν πυροβόλησαν ε, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες χρειάστηκε να απαντήσουν σε πυρά διακινητών. Οι διακινητές άνοιγαν πυρ και δυστυχώς υπήρξε ε, ένα θύμα, μια παράπλευρη απώλεια σε μία από αυτές τις ε, περιπτώσεις, σε ένα από αυτά τα επεισόδια το καλοκαίρι του 2015. Αυτά μπορώ να πω για αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, πυροβολισμών. Τώρα, τέθηκε μια ερώτηση για την σημερινή κατάσταση στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Σήμερα έχουμε περίπου 100 μετανάστες, 100-120 μετανάστες την ημέρα από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά. Το Φεβρουάριο τρέχοντος κατά μέσο όρο έφταναν από την Τουρκία στην Ελλάδα 2 με 2.500 άτομα το Φεβρουάριο δηλαδή συνολικά. Άρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Τα hot spot και χώροι υποδοχή για μετανάστες ε, στα ελληνικά νησιά είναι παρόλα αυτά σε πλήρη συμφόρηση. Ε, συνήθως ε, στεγάζονται διπλάσια από όσους θα έπρεπε να στεγάζονται από το δυναμικό η λειτουργία σε επιχειρησιακό επίπεδο με την Τουρκία, η συνεργασία με, το, με την Τουρκία σε επιχειρησιακό επίπεδο λειτουργεί. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι οι ακτοφύλακέ του κάνουν ενέργειε εντό των δικών του χωρικών υδάτων ε, διάσωση και για την ε, εφαρμογή της συμφωνίας επιστροφής μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία και τη δήλωση τη 20 η Μαρτίου οι τουρκικές αρχές έδειξαν πάντα πνεύμα συνεργασία σε επιχειρησιακό πλαίσιο όπως είχε συμφωνηθεί από το Συμβούλιο της Ένωσης και τι τουρκικέ αρχέ. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά για να απαντήσω σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που έχουν σχέση με τα σημεία επαφής στα τη μελη για να υπάρχει μηχανισμό προσφυγών. Το σκεπτικό είναι ότι εντός της υπηρεσίας ο αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ανεξάρτητος ε, από τον εκτελεστικό διευθυντή κατά την ε, διεξαγωγή ερευνών για καταγγελίες. Δηλαδή, όταν μέλη του προσωπικού από τις ε, χώρες που έχουν αναπτυχθεί υπό την αιγίδα επιχείρησης Frontex εμπλέκονται σε καταγγελόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει και οι εθνικές αρχές να ορίζουν κάποιον ε, μεσολαβητή ή κάτι τέτοιο, κάποιον ανεξάρτητο εν πάση περιπτώσει, για να είναι συνομιλητής του αρμοδίου θεμελιωδών δικαιωμάτων της Frontex για να γίνουν οι έρευνες στο εθνικό επίπεδο. Η Frontex θα οργανώσει μια συνάντηση με τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθεί αυτό ακριβώς το δίκτυο έχει προγραμματιστεί. Αν θυμάμαι καλά θα γίνει το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες και το αποτέλεσμα που αναμένουμε είναι τα κράτη-μέλη να ορίσουν συγκεκριμένους ε, ανεξάρτητους συνομιλητές έτσι ώστε να υπάρχει το δίκτυο για να προχωρήσουν αυτές οι έρευνες. Ε, όσον αφορά την πρόσβαση στο μηχανισμό προσφυγών, ναι, αν μπορούμε να το βελτιώσουμε θα το κάνουμε. Αλλά πρέπει να πω ότι στα hotspot και στις ε, κοινέ επιχειρήσεις και πριν από την ανάπτυξη των ε, δικών μας ανθρώπων υπάρχει μια εκπαίδευση έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συνοριοφύλακες ε, και οι εκτοφύλακες ε, τον μηχανισμό αυτών και πώς να αντιμετωπίσουν ε, μετανάστες άτομα που θέλουν να κάνουν κάποια καταγγελία. Μπορούν να το κάνουν είτε στη σελίδα είτε να τυπώσουν το έντυπο και να το κάνουν στο χαρτί. Για τις προσλήψεις και το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γιατί είχαμε ένα άτομο και τώρα έχουμε γραφείο έχουμε κάποιον υπεύθυνο δηλαδή συν ε, ένα άλλο άτομο που τον βοηθά για τις ε, προσλήψεις λοιπόν στις τρέχουσες προσλήψεις υπάρχουν κάποια άτομα που ασχολούνται με τις ε, καταγγελίες και σύμφωνα με τον αρμόδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη προσφυγή μέσω του νέου μηχανισμού αλλά βεβαίως έχουμε προγραμματίσει να προσλάβουμε τον Ιανουάριο γιατί εγώ είμαι και υπεύθυνο ε, και για την χρήση των πόρων. Ε, έδωσα το πράσινο φως στον αρμόδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα να εκδώσει μια προκήρυξη για την πρόσληψη δύο ατόμων και μόλις ο προπολογισμό του 17 εγκριθεί θα μπορεί η αρμόδια για τα θεμελιώδη δικαιώματα να προσλάβει τα άτομα αυτά. Για τις δεξαμενές από παντλούμε αυτή τη στιγμή προβλέπονται οι διάφορες δεξαμενές, ε, τρεις για τις επιστροφές, μία δεξαμενή προσωπικού ταχείας αντίδρασης για φυλακή και ακτοφυλακή. Έχουμε λοιπόν ε, την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρώσουμε την δημιουργία αυτών των δεξαμενών. Αυτό το οποίο θα έχουν τα κράτη-μέλη αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη είναι να διαθέσουν κάποιους ε, συνοριοφύλακες ε, και λιμενικούς ε, για την δεξαμενή ταχείας αντίδρασης. Κάθε κράτος μέλος ξέρει πόσους θα διαθέσει και θα μας πει. Είμαστε σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τους αριθμούς για το κάθε προφίλ, γιατί χοντρικά ο κανονισμός λέει πόσους, αλλά μετά πρέπει να δούμε τι είδους ανθρώπους θέλουμε. Παραδείγματος χάρη χώρες όπως να ε, πούμε στην κεντρική Ευρώπη, περίκλειστες χώρες, πιθανότατα δεν θα έχουν λιμενικούς. Οπότε δεν θα μας διαθέσουν. Οπότε εξαρτάται από τη γεωγραφία, από τις ανάγκες, αλλά οι συζητήσεις ε, είναι εν εξελίξη με τα κράτη-μέλη και αναμένω να οριστικοποιηθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου φέτος. Συνεργασία με τρίτες χώρες, ε, υπήρχαν πολλές ε, ερωτήσεις. Υπήρξε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις χώρες του δρόμου του μεταξιού που αναφέρθηκε, μια πρωτοβουλία δηλαδή με την οποία είχε συνδεθεί η Frontex ε, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για χώρες όπως το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν. Ε, για χώρες σε, αυτή την περιοχή του πλανήτη, εν πάση περιπτώσει. Οπότε για τι είδους συνεργασία έχουμε γενικώ με τρίτες χώρες. Έχουμε κάποιες ε, συνεννοήσεις, ε, διευθετήσεις, ε, συνεργασίας, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε περισσότερα τις λεπτομέρειες. Παραδείγματο χάρη με τις βαλκανικές χώρες και με χώρες υποψήφιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δυνητικά υποψήφιες. Η κατάσταση είναι διαφορετική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συνεννοήσει για να προετοιμάσουμε την ένταξη, να του τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν περισσότερες δυνατότητες, ε, να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τους ε, κανονισμού όσον αφορά την διαχείριση συνόρων ε, μετανάστευσης που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε άλλες χώρες ε, μακριά από την Ευρώπη οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προοπτική να γίνουν μια, χώρα, μια μέρα υποψήφιες χώρες οπωσδήποτε μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για την ανάλυση κινδύνου αλλά ε, δεν μιλάμε ε, βεβαίως για προσωπικά δεδομένα τι υπάρχουν κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων και είναι σαφές πως δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο. Για την επανεισδοχή. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Όρισα κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την εφαρμογή των συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κρατημέλη δηλαδή, μετά από την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η υπηρεσία ακολουθεί αυτά τα οποία γίνονται και σε επιχείρησεις επιστροφών, ισχύουν δηλαδή οι προδιαγραφές μας. Όσον αφορά την παρακολούθηση μπορώ να σας πω πως την εποπτεία Υπήρξαν πολλές φορές καταστάσεις που ανέφεραν ΜΚΟ ή βουλευτές όπου ε, ελέγχουμε. Σύμφωνα με τους κανόνες και τον κανονισμό και το ευρωπαϊκό δίκαιο η υπηρεσία δεν είναι αρμόδια για να αξιολογήσει το εάν η επιστροφή ενός ατόμου δικαιολογείται και δεν αποφασίζει. Η υπηρεσία όμως πρέπει να φροντίσει ότι υπάρχει η σωστή επιτήρηση και ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την επανεισδοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με ενημέρωσε μια γνωστή ΜΚΟ πριν από λίγες εβδομάδες και είπε ότι δύο άτομα θα επιστρέφονταν από την Ελλάδα στην Τουρκία και με ειδοποίησαν ότι υπήρχε μια απειλή και ότι ίσως τα άτομα αυτά θα διώκονταν ή ότι δεν αισθανόταν ε, ασφαλή εάν ε, επιστρέφονταν. Ε, δεν είναι στην εντολή αλλά αμέσως ήρθα σε επαφή με τις ελληνικές αρχές ε, ρώτησα για τα ονόματα αυτά, δεν ήταν στην λίστα της επομένης, οπότε τους ενημέρωσα ότι τα ονόματα αυτά δεν ήταν στη λίστα επιστροφών για την επόμενη επιστροφή. Υπήρξε επίσης μια περίπτωση πρόσφατα που αφορούσε ε, υπηκόους Συρίας που είπαν ότι δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα. Το ερευνούμε αυτό μαζί με τις ελληνικές αρχές, παρά το ότι και πάλι αυτό δεν είναι απολύτως εντός ε, της εντολής μου. γιατί βεβαίω πρέπει να σεβόμαστε τις ε, εθνικές αποφάσεις αλλά οπωσδήποτε οι πόροι που έχει η υπηρεσία δεν ε, χρησιμοποιούνται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά, ε, ξέρετε, από νομική σκοπιά είναι πολύ δύσκολο το θέμα και θέλουμε οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, με συγχωρείτε, λέει, ο πρόεδρος, οι διερμηνείς ε, πρέπει να αποχωρήσουν, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι μπορούν να συνεχίσουν στα αγγλικά. 12 και 35 αν δεν σας πειράζει. Γιατί ε, θέλουμε να ακούσουμε οπωσδήποτε τις απαντήσεις. Εντάξει Νάταλη, είπε, μπορείς να παρακολουθήσεις, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θέλω να ακούσουμε τις απαντήσεις, αλλά σήμερα οι διερμηνείς έχουν να πάνε και αλλού.